Περιμένουμε λίγο ακόμη. Περιμένουμε τον κύριο Μποβέ. Γιατί ήθελα να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα για την γεωργική πολιτική. Και παρόλα αυτά δεν έχει έρθει ακόμη. Ελπίζω να έρθει σε λίγο. Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, με θέματα προβλήματα της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2020 και το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Έχουμε κάνει την εισαγωγή. Το πιο σημαντικό είναι ότι παρίσταται ο κύριος Δόρφμαν που ήταν ακριβώς ο εισηγητής μας ε, ε, για την έκθεση αυτή, την ομώνυμη. Και μάλιστα πριν από λίγο ψηφίσαμε και όλα την έκθεση Ντόρφμαν. Με την ε, ακρόαση αυτή ε, θα βοηθήσουμε περαιτέρω τον εισηγητή Ντόρφμαν ενώπιση της Ολομέλειας και θα εμπλουτίσουμε και τη μελλοντική συζήτηση μετά την υποβολή και των νομοθετικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την μελέτη εκπώνησε το Ευρωπαϊκό, Περιβαλλοντικό, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε συνεργασία με μεμονωμένους ε, εμπειρογνώμονες από το Trinity College του Δουβλίνου, το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, το Reading University και το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας. Και τη μελέτη τη διαχειρίστηκε το Τμήμα Πολιτικής Β. Έχουμε και το χρονοδιάγραμμα που πάντα ε, μας πιέζει και διαρωτόμαστε αν θα τα καταφέρουμε να το τηρήσουμε ή όχι, αλλά έχουμε και πολλά ουσιαστικά ζητήματα που θα μας παρουσιάσουν οι εμπειρογνώμονές μας με τη δική τους άποψη, όχι μόνο την προσωπική τους άποψη, αλλά και την άποψη του επιτελείου τους, των συνεργατών τους. Μάλιστα μας έχουν στείλει και υλικό. Έχουμε την πλήρη δημοσίευση και μία σύνοψη. Όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε διάσταση απόψεων και ένα ευρύ φάσμα θέσεων για το θέμα αυτό. Έχουμε τον κύριο ε, Μπότερ Σχέντα από την ε, πολιτική Motorshead από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και τον κύριο Ζαν Κριστόφ Βιρό από το Μη Ιαπωνίας του Πανεπιστημίου του Παρισιού Σακλέ. Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για τη παρουσίαση που θα μας κάνουν και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Έχουμε μια μισή ώρα για τη συζήτηση. καθυστερήσαμε λίγο. Εμείς φταίμε γιατί περιμέναμε περισσότερους ευρωβουλευτές. Έχετε 15-20 λεπτά για την παρουσίαση, κύριε Μότερσετ. Παρακαλώ. Uh, actually, Mr. Chairman... Κύριε Πρόεδρε, ε, η παρουσίαση είναι κοινή και των δυο μας. Ως εκ τούτου δεν θα χρειαστούμε και οι δυο, και δύο μαζί 20 λεπτά, άρα θα παραμείνει αρκετός χρόνος για συζήτηση. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, η υπηρεσία Quick μας ε, ανέθεσε να σχολιάσουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση λοιπόν που έχετε μπροστά σας, ε, πρέπει να το υπογραμμίσω, είναι ένα σχέδιο. Η έκθεση αυτή είναι ευσύνοπτη, θα ακολουθήσει μία μακροσκελέστερη έκθεση, απλά αυτή η έκθεση είναι προς ενημέρωση και θα ακολουθήσει μία, όπως σας είπα, μακροσκελέστερη έκθεση όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη μετά από μία μισή περίπου εβδομάδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σύντομα θα σας παρουσιάσω την ομάδα της μελέτης, το αντικείμενο της μελέτης και πώς ακριβώς εντάσσεται στα πολιτικά ορόσημα, όπως τα λέμε, της μεταρρύθμισης της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Να δούμε τι είναι το καινούργιο στην ανακοίνωση της Κομισιόν, πώς τα αναλύουμε αυτά και πώς όλες αυτές οι απόψεις μπορούν να δραματίσουν ε, κάποιο ρόλο στην νομοθετική διαδικασία. Ποιοι είμαστε? Είμαστε το Ινστιτούτο για Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική. Είναι μια ε, δεξαμενή ε, Σκέψει και Εγκεφάλων που συνεργάζεται και με την κοινωνία των πολιτών και με ΜΚΟ αλλά και με ιδιώτες. Ε, διεξάγουμε έρευνες ε, η μελέτη λοιπόν αυτή, στην οποία συμμετείχαν και ο καθηγητής κ. Πύρου και ο κ. Μάθιους και οι δύο είναι διακεκριμένοι οικονομολόγοι που ασχολούνται με θέματα γεωργίας και φαντάζομαι θα γνωρίζετε τις ε, εργασίες τους. Αυτό που μας ζητήθηκε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε την ε, ανακοίνωση, να τη συγκρίνουμε με τους στόχους ε, που έχουν τοθεί και επίσης να δούμε και τι άλλο κυκλοφορεί, ε, να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ε, συστάσεις. Η έκθεση δεν θα ήταν ενδιαφέρουσα αν δεν βλέπαμε τη διατύπωση στην ανακοίνωση που είναι σε κάποιες περιπτώσεις ε, αρκετά συνοπτική, άρα δηλαδή λάβαμε υπόψη μας πάρα πολλές απόψεις όπως ακριβώς προέκυψαν από συζητήσεις και σεμινάρια και άλλες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι αυτοί προσπάθησαν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, ακόμα και αν σε αυτή τη φάση της διαδικασίας τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Ε, όσον αφορά το πολιτικό περίγραμμα, πολλοί θα έχετε διαπιστώσει ότι εκεί εντάσσονται οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα λάβουν χώρα το Μάιο του επόμενου έτους. Είναι λοιπόν λιγάκι δύσκολο να διαβλέψουμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα επανέλθουμε αργότερα στις συστάσεις μας επ' αυτού. Περνάμε στην ίδια την ε, ανακοίνωση ε, να δούμε λιγάκι τι ακριβώς περιλαμβάνει. Πρόκειται για τον συνδυασμό ε, στόχων ε, για το ότι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων έχει γίνει πλέον σήμερα ένα απόλυτα συνδυασμένο στοιχείο με τις ισορροπίες οι οποίες περιγράφονται ως ε, η ενίσχυση του κοινωνικονομικού ιστού. Ε, θα μου επιτρέψετε να δώσω και κάποια στοιχεία σχετικά με το που αποδίδει σημασία αυτή η πολιτική. Η πολιτική, η βιώσιμη, ε, συνεπάγεται ότι θα υπάρχει ένας μεγαλύτερος ρόλος της πολιτικής και επίσης και η συμπεριφορά των γεωργών και αυτή θα είναι καθοριστική σημασία. Όσον αφορά το δεύτερο βασικό στοιχείο που προκύπτει από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σχέση με την πρόταση για μαζική ενίσχυση της επικουρικότητας. Να αναλάβουν περισσότερες αμμοδιές στα κράτη-μέλη που θα κληθούν όχι μόνο να καταρτήσουν νέες, στρατηγικά σχέδια για το σύνολο της κοινή γεωρικής πολιτικής, αλλά τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν και τον σχεδιασμό και τον έλεγχο πολλών από τα ίδια τα μέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχολιαστεί αρκετά στις ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν στην έκθεση. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον Ζαν Κριστόφ, ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει την ε, γεωργία αντοχής. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επιτύχει αυτή την ευφυή και ανθεκτική γεωργία. Υπάρχουν ε, αρκετά στοιχεία στην ανακοίνωση ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, καλύτερη στόχευση των άμεσων ενισχύσεων. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες προτάσεις για περιορισμό αυτών των ενισχύσεων. Υπάρχει εξάλλου και η πρόταση ότι οι μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες πραγματικά ασχολούνται με τη γεωργία θα πρέπει να αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο και κάποιες άλλες απόψεις ότι επειδή είναι απαραίτητο να υπάρχει ανανέωση των γενεών ε, θα πρέπει να γίνονται ίσως ε, καταβάλλονται περισσότερες ενισχύσεις στους νέους γεωργούς ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημασία αποδίδεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό αναφέρεται επανειλημμένα στην έκθεση και αναγνωρίζεται ότι ρόλο παίζει το επίπεδο της εκπαίδευσης των γεωργών που ποικίλει ανάλογα με το κράτος. Ε, στο τέλος της έκθεσής μας εμείς αναφέρουμε διάφορα στοιχεία και εκεί εντυπωσιάζουν πραγματικά οι διαφορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι οι πολιτικές ε, δεν αποσκοπούν ε, στο ανθρώπινο κεφάλαιο ή δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Κυρίως όσον αφορά το σύστημα παροχής γνώσεων και πληροφοριών. Υπάρχουν αντικείες και αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αναφέρεται επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν και περαιτέρω προσπάθειες έτσι ώστε οι γεωργοί να έχουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην αλυσίδα της αξίας μέσα από συμμετοχή σε περισσότερες διαπραγματεύσεις. Επ' αυτού δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες αλλά θα ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες σχετικά με την οδηγία για αθέμητες εμπορικές πρακτικές τι είναι η ανάλυση αυτών των ε, θεμάτων. Υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσον η ανακοίνωση πράγματι επιτυγχάνει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη του εισοδήματος αφενός ε, με ε, καταβολή άμεσων ισχύσεων χωρίς διακρίσεις που να επηρεάζουν θετικά το εισόδημα. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες αυτό. Αυτό είναι το ένα και από την άλλη υπάρχουν οι επενδύσεις για την βελτίωση της ε, παραγωγικότητας. Η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε κάποιο βαθμό ε, είναι και απογοητευτική όσον αφορά την απόδοση, όσον αφορά την παραγωγικότητα, των συντελεστή παραγωγικότητας ε, που και αυτός ε, δεν είναι ενθαρρυντικός ε, γιατί συνδυάζεται και με τη μείωση της απασχόλησης στη γεωργία. Τίθεται και το ερώτημα κατά πόσον όλες αυτές οι επενδύσεις στην κοινή γεωργική πολιτική τις τελευταίες δεκαετίας μήπως θα ήταν καλύτερα να έχουν τοποθετηθεί στο να βελτιωθεί η απόδοση της γεωργίας. Αυτό προκύπτει και ως ερώτημα μετά την ανακοίνωση. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι η ανακοίνωση ενθαρρύνει την είσοδο νέων γεωργών στη γεωργία, αλλά πρέπει να πω ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προτάσεις που να προχωρούν πιο πολύ από αυτά που ήδη προβλέπει ο κανονισμός του 2013. Δηλαδή ε, και συνεργασίες για καινοτομία που αφορούν στη γεωργία. Γενικά υπάρχουν θετικές αξιολογίες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο οποίο τα κράτη-μέλη προσεγγίζουν το θέμα. Υπάρχει ε, κάποια ανισότητα στο θέμα αυτό. Εξάλλου, ε, σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει απόλυτη συμμετοχή γιατί είναι πολύ λίγοι οι γεωργοί ε, οι οποίοι συμμετέχουν στην λειτουργική ομάδα. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε περισσότερο παρότι τα εργαλεία ήδη περιλαμβάνονται στην ε, σχεδιαζόμενη πολιτική. Υπάρχει λοιπόν μια άποψη η οποία έχει κατατεθεί από διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου ε, ότι οι συμβουλές που παρέχονται δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητες παραδείγματος χάρη από τους προμηθευτές σε ορισμένα κράτη-μέλη. Πρέπει να ε, το υπογραμμίσουμε ότι αυτό το σύστημα ενημέρωσης είναι συμβουλευτικό. Πώς προτείνει η Κομισιόν να ενισχύσει τον κοινωνικο-οικονομικό ιστό. Ε, προβλέπονται πρωτοβουλίες όπως ο καλύτερος συντονισμός, η άποψη ότι ε, θα πρέπει στο πλαίσιο της καλύτερης πολιτικής να εξετάζονται και πραγματικές επιπτώσεις στις ε, γεωργικές περιφέρειες. Υπάρχει και άποψη να συνδεθούν μεταξύ τους τα μικρά χωριά. Και όπως ήδη είπα υπάρχει και άποψη ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ανανέωση των γενεών για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της γεωργίας. Εξάλλου, η ανακοίνωση ε, υπογραμμίζει το ότι πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπιστεί το θέμα των κινδύνων και των διακυμάνσεων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανθεκτικότητα. Ε, αν αναλύσει κανείς τα θέματα, καταλήγει στο ότι η διασύνδεση προφανώς και βρίσκεται στον πυρήνα πολλών προτάσεων. Ε, η διασύνδεση είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και καλή σχέση ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή γεωρική πολιτική και το Ταμείο Συνοχής. Υπάρχει και μια πρόταση να συνδεθούν μεταξύ τους τα διάφορα μικρά χωριά, αλλά να υπάρχουν ε, και στοιχεία έτσι ώστε να λειτουργήσει αυτός ο νέος μηχανισμός και για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να ε, συγκεντρωθούν δεδομένα. Απαραίτητο επίσης ε, να πλουστευτεί και η κοινή γεωργική πολιτική. Εξάλλου η διασύνδεση είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε καλύτερη απόδοση ε, της συμβουλευτικής υπηρεσίας για τη γεωργία που έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη γενικότερη απόδοση της γεωργίας. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι νέοι γεωργοί ε, αποτελούν κεφάλαιο για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Είναι όμως επίσης απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση. Όταν θα αποσύρεται ένας ε, ηλικιωμένος ε, γεωργός, ε, όχι απαραίτητα να τον διαδέχεται ο γιος του ή η κόρη του, πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένα τα παιδιά και γι' αυτό έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος αυτού. Υπάρχει μια δυνατότητα να συνδέσουμε τις ενισχύσεις ε, για εκπαίδευση και συμβουλές ε, ε, σε όλο αυτό το μηχανισμό που προανέφερα. Βεβαίως το επίπεδο εκπαίδευσης των εισερχόμενων είναι καθοριστική σημασίας και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Όσον αφορά τους κινδύνους και τις διακυμάνσεις των εισοδημάτων, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση Νομίζω αυτό πρέπει να το στηρίξουμε και υπάρχει και η ιδέα του να βασιστούμε περισσότερο στην ανθεκτικότητα, στην αντοχή των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κάποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν ε, τα σοκ από τη διακυμάνση των ε, τιμών. Ε, αυτό αφορά εκείνες τις εκμεταλλεύσεις που τους, λόγω του χαμηλού κόστους μπόρεσαν να απορροφήσουν τους κραδασμούς η διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να συνδέεται και με την μετάβαση προς μια τέτοια μορφή γεωργίας που θα είναι περισσότερο βιώσιμη και θα εξαρτάται περισσότερο από τις ε, αγορές και τις εισρωές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στις φιλοδοξίε της Κομισιόν σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Λέμε ξεκάθαρα πως Είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι στο παρελθόν, αλλά είναι δύσκολο βεβαίω να το δει κανείς. Στο διάγραμμα εδώ στα αριστερά βλέπετε την υφιστάμενη πράσινη αρχιτεκτονική της με την πολλαπλή συμμόρφωση στο κάτω μέρος. Το πρασίνισμα, το λεγόμενο. Οπότε Βλέπετε την ε, τωρινή πράσινη αρχιτεκτονική όπου έχουμε την πολλαπλή συμμόρφωση, το πρασίνισμα και τα κλιματικά περιβαλλοντικά μέτρα. Στα δεξιά βλέπετε ένα αρκετά καθησυχαστικό διάγραμμα που δείχνει πως έχει απλοποιηθεί η πολλαπλή συμμόρφωση και το πρασίνισμα σε μια νέα ενισχυμένη αίρεσιμότητα που είναι κάπως πιο φιλόδοξη γιατί το κουτί, αν το δείτε, φτάνει κάπως λίγο πιο ψηλά και υπάρχουν μετά τα μέτρα του πυλώνα 2 επιπλέον αυτού, συν μια πρόταση για ένα εθελοντικό περιβαλλοντικό σχέδιο στον πυλώνα 1. Οπότε η Κομισιόν παρουσιάζει μια εικόνα ότι θέλει δηλαδή να επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντική φιλοδοξίας ε, στον πυλώνα 1 και 2. Πρέπει βεβαίω να το δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό ε, λεπτομέρειας. Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε ακόμα είναι το πώς η νέα αυτή ενισχυμένη αίρεσιμότητα που σημαίνει δηλαδή το πρασίνισμα και η πολλαπλή σε ένα μέτρο πώς θα αυξήσει την λεγόμενη φιλοδοξία. Και το σημαντικότερο θα ανησυχούσαμε αν λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η πολλαπλή συμμόρφωση. Γιατί αυτές οι απαιτήσει δίνουν τεράστια διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη αυτή την στιγμή και βλέπουμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα σε αυτά τα οποία κάνουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ένα χωράφι με κλίση 7 βαθμούς θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα μέχρι να διπλασιαστούν οι ε, μοίρες της κλίσης. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι ε, πρέπει να υπάρχει ένας κοινό πύρινας ε, της ενισχυμένης αιρεσιμότητας και μία από τις τροπολογίες στην έκθεση του κυρίου Ντόρφμαν μιλάει για αυτό ακριβώς το πράγμα. Ένα κοινό πυρήνα δηλαδή που θα επηρεάζει όλους τους αγρότες. Αναφέραμε τα οικολογικά σχέδια στον πυλώνα 1 αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πως είναι εθελοντικό και δεν αντικαθιστά τον πολύ σημαντικό συμβολισμό του 30% που πηγαίνει στο πρασίνισμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να τα δούμε αυτά στο πλαίσιο του πι για να υπάρξει μια περιχαράκωση της χρηματοδότησης αυτής και να μην υπάρχει υποβάθμιση από το 30% που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το πιο ριζοσπαστικό θέμα εδώ με τις νέες προτάσεις είναι ο νέος μηχανισμός ε, υλοποίησης. Θεωρούμε ότι το σκεπτικό αυτό, ότι δηλαδή ολόκληρη η ΚΑΠ θα πρέπει να συνεισφέρει σε κάποιους στρατηγικούς στόχους, είναι κάτι το θετικό. Θα μπορούσε ο πυλώνας 1 να χρησιμοποιείται με πιο στρατηγικό τρόπο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Γιατί μέχρι τώρα το πρασίνισμα χρησιμεύει για πράγματα τα οποία είναι βολικά για τις διοικήσεις και απλά για τους αγρότες, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν με τρόπο στρατηγικό, ακόμα και με τα μέτρα που βρίσκονται τώρα στον πυλώνα 1. αλλά δεν μπορούμε να τονίσουμε το πόσο δύσκολο θα είναι να ξεκινήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για διάφορους λόγους. Το ένα είναι η δυνατότητα και η πολιτική βούληση να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμό όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά χρημάτων, όταν ο κόσμος έχει ε, μια συγκεκριμένη εμπειρία από την ΚΑΠ ε, και δεν ξέρω αν θα έπρεπε κάποιος να ε, σκεφτεί πως να κρατήσουμε το παλιό σύστημα μέχρι να μάθει ο κόσμος ε, το καινούριο. Ένα άλλο εμπόδιο είναι ο σχεδιασμός του πι Αν έχουμε δηλαδή κάποια μέτρα που δεν συγχρηματοδοτούνται, ενώ άλλα συγχρηματοδοτούνται, αντικειμενικά είναι δύσκολο να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Ανησυχούμε δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να κάνουν κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με ένα διαφορετικό περιβάλλον συγχρηματοδότησης. Υπάρχουν και κάποια τεχνικά εμπόδια, δηλαδή να κρίνουμε ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος, όταν κάποιος προσπαθεί να καθορίσει την εφαρμογή της κάποια το ποιοι θα είναι οι στόχοι, πώς μπορούν να μεταφραστούν σε δεδομένα μετρήσιμα θα είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και βεβαίως οι παράγοντες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ευνοούν το status quo. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν τα σχέδια αυτά εγκαίρως για να πληρωθούν οι αγρότες οι οποίοι δικαίως αναμένουν κάποια πληρωμή, υπάρχουν σοβαροί χρονικοί περιορισμοί για το πώς μπορεί να γίνει ένας ολιστικός στρατηγικός σχεδιασμός. Ναι, τελειώνω. Τα συμπεράσματά μας λοιπόν και οι συστάσεις μας θεωρούμε ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στις άμεσες πληρωμές, έστω και αν είναι πιο εστιασμένες. Θέλουμε να δοθεί περισσότερη έμφαση στο πώς ξοδεύονται τα χρήματα της χειρουργικής πολιτικής για να αυξηθεί η βιωσιμότητα και η αηφορία. Επίσης υπάρχουν μηχανισμοί που δημιουργούν στρεβλώσεις και αφορούν και αφορούν περισσότερο πράγματα, όπως οι συνδεδεμένες πλήρωμες. Αυτό θα πω μόνο. Και όπως είπα η Κομισιόν πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι υπάρχει σε αυτήν την νέα περιβαλλοντική αρχιτεκτονική. Τελευταία σελίδα, όπως είπα. Ο νέος μηχανισμός αυτός ε, απόδοσης ε, χρειάζεται, όπως σας είπα, νέα δεδομένα, δυνατότητες υλοποίησης από την πλευρά των κρατών μελών και πλησιάζουν και οι ευρωεκλογέ σε ένα χρόνο. Ίσως θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την περίοδο για να ε, υλοποιήσουμε κάποιες ιδέες πιλωτικά για να έχουμε μια πιο στερή νομοθετική διαδικασία. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ δηλώστε όσοι θέλετε το λόγο στη συζήτηση για να καταρτήσουμε κατάλογο αγορητών και να δούμε πως πώς θα κατανείμουμε το χρόνο. Ο κύριος Ντόρφαν πρώτος. Ε, μόνο στον κύριο Ντόρφμαν δεν θα περιορίσω το χρόνο αγόρευσης. Και παρακαλώ όσοι άλλοι θέλετε το λόγο να το δηλώσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα που ετέθησαν και νομίζω ότι τα θέματα αυτά τα ρυθμίσαμε στην έκθεση την οποία ψηφίσαμε σήμερα το πρωί. Κυρίως εκεί όπου γίνεται λόγος για τους νεοεισερχόμενους στη Γεωργία. Και έχω ένα ερώτημα. Εσείς περιοριστήκατε στον πρώτο πυλώνα. Νομίζω λοιπόν ότι όταν πρόκειται για την προθυμία νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη γεωργία. Στην περίπτωση αυτή, ε, καθοριστική σημασία είναι και ο δεύτερος πυλώνας. Δηλαδή, οι νέοι αυτοί άνθρωποι χρειάζονται ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο να μπορούν να διαβιούν μαζί με τις οικογένειές τους. Ρόλο δεν παίζει μόνο το οικονομικό στοιχείο, η απόδοση της ε, γεωργικής εκπετάλευσης. Προφανώς και αυτή είναι καθοριστική σημασία, αλλά δεν είναι το μόνο. Στην αξιολόγηση του New Delivery Model το οποίο παρουσιάσατε εσείς, ε, δεν άκουσα ακριβώς τη δική σας την άποψη. Δηλαδή, στη δική μου την έκθεση εκφράσαμε πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά στις στρεβλώσεις της αγοράς. Ε, ε οι στρεβλώσεις της αγοράς ε, είναι άμεσα συνδεδεμένες και με τις συνδεδεμένες πληρωμές, αλλά στρεβλώσεις της αγοράς μπορούν να προκύψουν και από πολλές άλλες αποφάσεις, όταν δηλαδή τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται τα κονδύλια που τους έχουν διαχειριστεί ε, σχεδόν απόλυτα κατά το δοκούν. Και εκεί ξεπερνούν τις συνδεδεμένες πληρωμές. Όσον αφορά το πράσινο οικοδόμημα ή αρχιτεκτόνημα, εγώ ε, αν κατάλαβα καλά, εσείς ε, ε, την ανακοίνωση της Κομισιόν ε, δεν τη βρίσκετε τόσο αρνητική. πρόκειται για λογική και ενισχυμένη αιρεσιμότητα στον πρώτο πυλώνα και λέτε ότι στον δεύτερο πυλώνα έχει κάθε νόημα να υπάρξουν προαιρετικά προγράμματα υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγκαστούν τα κράτη-μέλη στο δεύτερο πυλώνα να εφαρμόζουν και περιβαλλοντικά προγράμματα. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό που δεν συζητείται κατ' ουσίαν είναι το κατά πόσο αυτά τα προαιρετικά ε, εθελοντικά προγράμματα επικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό με τα προγράμματα του πρώτου πυλώνα. Στο πρασίνισμα το βιώσαμε αυτό. Ε, τα προγράμματα αυτά περιορίστηκαν στο δεύτερο πυλώνα γιατί υπήρχε κάποια αντίφαση με το πρασίνισμα. Δηλαδή ορισμένα μέτρα δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν στο δεύτερο πυλώνα ε, γιατί απλά ε, επικαλύπτονται απόλυτα με το πρασίνισμα και άρα δεν είχαν και κανένα νόημα. Κατά τα άλλα δεν είπατε εσείς τίποτα για τις αγορές των γεωργικών προϊόντων. Κατά την άποψή μου αυτό το θέμα των αγορών είναι καθοριστική σημασία. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για προαγωγή του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Πρέπει και να συζητήσουμε το πώς μια γεωργική πολιτική μπορεί να οργανώσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις αγορές και πώς ε, με τον τρόπο αυτό οι γεωργοί ε, θα προσπορίζονται το βέλτιστο, το υψηλότερο δυνατό εισόδημα από την πώληση των προϊόντων του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουαζό τώρα, για 1,5 λεπτό όμως. Πολύ λίγο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ τους ε, καταπληκτικούς ομιλητές μας. Κόντεψα να κοιμηθώ. Μάλιστα ένας Γάλλος που τόλμησε να μιλήσει αγγλικά. Ε, σας ε, υπενθυμίζω ότι η Γαλλία είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μαζί με τη Γερμανία. Γιατί μιλήσατε άλλη γλώσσα. Επίσης, ε, ε, έχουμε υποστεί πολλά από την ΚΑΠ και πριν σκεφτούμε τον οικολογικό προσανατολισμό, την ευφυή γεωργία, τους ε, κοινοτικούς δείκτες, γιατί δεν επαρερχόμαστε ε, στο θεμέλιο της ΚΑΠ, που είναι οι αγρότες. Οι αγρότες θα πρέπει να είναι η καρδιά της ΚΑΠ και όχι ο στόχος ή το θύμα της ΚΑΠ. Ε, οι αγρότες μας πουλούν ε, σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής. Οπότε θα πρέπει να αναδείξουμε τα προϊόντα, να προσπίσουμε τις γεωργικές ενδείξεις, ε, να σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών έχοντας κοινού στόχους και η επαναθηνικοποίηση της ΚΑΠ δεν είναι βρισιά. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην κοινή λογική και οι ευρωβουλευτές και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, γεωργία πριν την ε, γεωργική εκμετάλλευση. Το γεωργικό εισόδημα πριν ε, να προέχει του εισοδήματο των μεγάλων ε, βιομηχανιών. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες να λαμβάνονται πρώτα υπόψη πριν από τους μετανάστες μειώνεται ο πυλώνα, αλλά διακυβεύεται η επικουρικότητα. Θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη για μια καλύτερη προσαρμογή στι ε, τοπικέ Ευχαριστώ. Κύριο Κολομπιέ. Ή μήπως όχι. Δεν χρειάζεται. Η μήπω οχι Ζωανά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ε, τους καλεσμένους μας για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν, τους εμπειρογνώμονες. Η κοινή γεωργική πολιτική υποτίθεται ότι εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες ε, ώστε να απασχολούνται οι γεωργοί και να επιτελούν το έργο τους, στην παραγωγή τροφίμων δηλαδή. Ε, έγιναν κάποιες βελτιώσεις χάρη στην ΚΑΠ. Η παγκοσμιοποίηση όμως, ε, η οικονομική κρίση και οι κλιματικές αλλαγές μας υποχρεώνουν να καταρτήσουμε προτεραιότητες ως προς τους στόχους μας. Και ο γεωρικός προϋπολογισμός θα πρέπει τουλάχιστον να παραμείνει στα τωρινά επίπεδα. Θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους οι γεωργοί και να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Και χρειαζόμαστε πιο ελαστικούς στόχους στη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Νωρίτερα αναφερθήκατε στα ανώτατα όρια. Δεν νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με αυτά. Εγώ προτιμώ τα εθελοντικά ανώτατα όρια. Επίσης μας μιλήσατε για το δεύτερο πυλώνα. Θεωρώ ότι ο δεύτερος πυλώνας έχει σημαντικό ρόλο και μιλήσατε και για τις άμεσες για τις άμεσες ενισχύσεις που επίσης παίζουν κρίσιμο ρόλο και θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες, το πρόγραμμα είναι αρκετά καλό. Υπάρχει όμως μια διάταξη που κατά τη γνώμη μου πρέπει να διαγραφεί. Η διάταξη αυτή προπρέπει τη δυνατότητα ε, ε, της θέσπισης ε, ε επιδοτήσεων για τις ε, συντάξεις. Ε, θα πρέπει να διαγραφεί η διάταξη που αποτρέπει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέου γεωργού και να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε προποθέσει για να ασχοληθούν με τη γεωργία, αλλά ας μην ξεχνούμε τα, δι... κεκτημένα δικαιώματα των αγροτών που μπορεί να έχουν και άλλε δραστηριότητε. Δεν θα πρέπει να εκδιώξουμε τους συνταξιούχου από την Ήπεθρο. Χάρη στους αγρότες μας έχουμε ασφαλή υγιεινά τρόφιμα σε προσιτές τιμές στο τραπέζι μας και φυσικά και ποιοτικά τρόφιμα. Πώς μπορεί ένας γεωργός ε, να παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες χωρίς συστηματική χρηματοδοτική ενίσχυση. Ευχαριστώ κύριο Σάγνιο. Well, not surprisingly, Chairman, Θα σας προξενήσει η εντύπωση πως ε, με ενδιαφέρουν αυτές οι λέξεις ε, κλιματική δράση. Τι θα είναι αυτή δηλαδή. Είναι μείωση στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου λιγότερο διοξείδιο του ανθρακάνων ναι, θα μπορούσαν να το μειώσουν οι αγρότες εάν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γλυφοσάτη και γενετικά τροποποιημένα φυτά. Το ίδιο και με το μεθάνιο, με το να μειώσουν τα μυρικαστικά, μετά αζωτούχα οξύδια. Να, πώς γίνεται αυτό, να σταματήσουν να καλλιεργούν ψυχανθή. Τι τους λέει όμω η Κομισιόν, α όχι, όχι, περισσότερα πρωτεϊνούχα φυτά. Οπότε εδώ πέρα έχουμε κάποιες σοβαρέ αντιφάσει. Τι σημαίνει λοιπόν τελικά κλιματική δράση. Τώρα όσον αφορά τις νέες πληρωμές για νέες δράσεις, εγώ θα ήθελα να μπορούν να φύγουν οι ηλικιωμένοι αγρότες με αξιοπρέπεια και να μπουν νέοι αγρότες στη δουλειά καλό είναι να μην τους δίνουμε λεφτά αλλά εγγυήσει δανείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μετρητά στην υποδομή βιοασφάλειας. Αυτοί οι αγρότες που έχουν βιοασφάλεια και σχετικές υποδομές υποφέρουν λιγότερο από ασθενείς. Θα ήθελα επίσης να υπάρξει κάποια χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά εκείνα σχέδια τα οποία κάνει από μόνος του ο κλάδος. Παραδείγματος χάρη να έχουμε τα ζαχαρότευτλα και τα όριζα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μελέτη, αλλά αυτό που μου λείπει είναι ότι δεν κατάλαβα ποια είναι η δική σας η θέση. Δηλαδή, ε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, τελικά υπάρχει κάποιο όρομα, ε, υπάρχει ένα κίνητρο για να προκύψει συζήτηση και Λόγω του ότι μέχρι τώρα η κοινή γεωρική πολιτική δεν τα πάει και πολύ καλά όσον αφορά τη βιωσιμότητα, εγώ προσωπικά διαρωτώ με ως έχουν τα πράγματα, ε, ίσως θα πρέπει να υπάρξουν ε, περικοπές στον πρώτο, μετά και στον δεύτερο πυλώνα και κατά πόσον με αυτές τις περικοπές μπορούμε να έχουμε ε, μια πραγματική οικονομική καλή απόδοση. Ειδικά σελίδα 8, αναφέρομαι σελίδα αυτή, εκεί εσείς ε, λέτε με σαφήνεια ότι χρειαζόμαστε αύξηση της ε, παραγωγής, ε, λύση λέτε είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, όμως αυτό αντιφάσκει με όλη αυτή την άποψη περί προστασίας του περιβάλλοντος. Φοβάμαι ότι σε αυτά που μας είπατε υπάρχουν αρκετά κενά, κυρίως στη σελίδα υπαριθμών 11 εκεί εσείς παρουσιάζετε μόνο το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν υπάρχουν παραδείγματα από εσά για το τι μπορούμε να βελτιώσουμε για μένα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα ανοιχτά ερωτήματα από λύσεις που θα μπορούσα να πω ότι μας προτείνατε. Ε, δεν νομίζω ότι με αυτά που μας είπατε καταλήγουμε στο ότι πράγματι υπάρχει μια καλύτερη βάση πάνω στην οποία να συζητήσουμε. Thank you, um, Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ και ευχαριστούμε τους ε, εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση. Εγώ θα σταθώ σε μία σύστασή σα ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στι άμεσε ενισχύσει. Και υπάρχει και το πρόβλημα τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτό όμω ε, αντιβαίνει σε πολλά μηνύματα που ε, παίρνουν οι γεωργοί από του ε, οικολόγου. Ότι είναι υπερβολικά εντατική δηλαδή η γεωργία. Και υπάρχει και μία αντίφαση σε αυτά που μα παρουσιάσετε και εσεί. Επίση, αν είναι κανεί αγρότη και εξαρτάται απόλυτα από τι άμεσε ενισχύσει για το γεωργικό του εισόδημα, ε, φυσικά και θα πρέπει να δώσει έμφαση για το εισόδημά του που ε, μιλάμε, για το βιο, βιοπορισμό του. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο και της παρουσίασης. Και το πρωί ψηφίσαμε για ένα νέο πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών ε, που θα, θα απομακρύνεται από τα ιστορικά δικαιώματα. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και ναι, μεν είναι καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να την επεξεργαστούμε και να δούμε πώ θα λειτουργήσει σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευση και πώ θα κατανεμηθούν τα κονδύλια. Επίση, το θέμα τη κατάρτιση των νέων αγροτών. Αυτό στην Ιρλανδία είναι τμήμα του πακέτου, δηλαδή θα πρέπει κανεί να ακολουθήσει κατάρτιση για να δικαιούται κονδύλια. Και με εντυπωσίασε, με εξέπληξε το σχόλιο σα για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δεκάστρο, καθηγητή Δεκάστρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και του συναντέλφου για αυτά που ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μόνο μία ερώτηση, ξεκάθαρη ερώτηση. Αυτό ε, το στοιχείο που λέτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιδεικνύουν κάποια ευελιξία όσον αφορά το νέο μοντέλο απόδοσης, New Delivery Model. Δεν θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα στα κράτη-μέλη, κυρίως εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία εκ του συντάγματος διαδραματίζουν ρόλο και σε μεμονωμένες περιοχές. Ε, αναφέρομαι στο κατά πόσον υπάρχει αυτονομία στην γεωρική πολιτική αφορά την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία. Δηλαδή τελικά με όλα αυτά δεν υπάρχει ο κίνδυνος ε, να προκύψουν περισσότερες τρευλώσεις από αυτό το νέο μοντέλο. Ε, περισσότερες από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα από τα εφαρμοζόμενα σχέδια ανάπτυξης. Επίσης υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος, το κίνδυνο συγχρηματοδότησης ε, στον πρώτο πυλώνα. Ε, αν κάθε περιοχή κάνει δύο σχέδια, ένα για τον πρώτο και ένα σχέδιο για το δεύτερο πυλώνα, γιατί τότε η περιφέρεια να μην τα χρηματοδοτεί όλα το να αφήνει κανείς την αυτονομία πλήρως ε, στα χέρια των κρατών μελών. Εσείς δεν πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για την κοινή γεωργική πολιτική. Δηλαδή η κοινή γεωργική πολιτική πράγματι κινδυνεύει να γίνει πλήρως επανεθνικοποιημένη. Κύριος Βάιτς. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Έχω τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπατε για στρεβλώσεις της αγοράς αν υπάρξουν επανεθνικοποίησεις. Το ερώτημά μου είναι ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες που πρέπει να παραμείνουν οπωσδήποτε κοινέ. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την παρέμβαση στην αγορά. Πώς βλέπετε δηλαδή την παρέμβαση σε κάποια τμήματα της αγοράς έτσι ώστε η προσφορά να συμφωνήσει με την ε, ζήτηση έτσι ώστε να γίνουν και οι αγρότες κάπως πιο ανεξάρτητοι από τις εξελίξεις της αγοράς. Και τέλος, πώς βλέπετε γενικώ ε, την άποψη ότι θα πρέπει να δίνονται στρεματικές ενισχύσεις μόνο εάν πληρούνται όλοι οι όροι οι περιβαλλοντικοί και της ε, υγιεινής των τροφίμων. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτά που ακούσαμε από τους καλεσμένους μας και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Ελπίζω όμως να είστε λίγο πιο σαφείς στις απαντήσεις. Πιστεύετε ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βελτιώσει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία ή θα την επιδεινώσει. Γιατί θα μειωθούν λόγω του Brexit τα γεωργικά κονδύλια. Και ήδη έχουν δημοσιευθεί κάποια στοιχεία αριθμητικά που δείχνουν αρκετή μείωση του γεωργικού προπολογισμού. Σχετικά υψηλό ποσοστό μείωσης. Επίσης, οι νέοι δεν, προσελ... δεν ελκύονται από τη γεωργία, προτιμούν άλλα επαγγέλματα. Δεν είναι πια ελκυστική η γεωργία. Και στην πατρίδα μου, τη Λιθουανία και γενικώ στις χώρες της Βαλτικής, οι αγρότες μας προτιμούν να αποδημούν σε άλλες χώρες για να ασχοληθούν με τη γεωργία, γιατί είναι τέτοιες οι διακοιμάνσεις των τιμών και οι και η αστάθεια του εισοδήματος που είναι πολύ αποκαρδιωτικές για τους γεωργούς που προσπαθούν να αναζητήσουν καλύτερο μέλλον σε άλλη χώρα. Επίσης υπάρχουν ανισορροπίες στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων και τα κονδύλια ε, που χρηματοδοτούν ε, τους γαλακτοπαραγωγούς ε, πηγαίνουν προς τους λιανεμπόρους που μειώνουν τις τιμές χωρίς μηχανισμό ρυθμιστικό και διορθωτικό. Τι έχετε να πείτε για αυτό το στοιχείο. Επίσης, θα καταφέρουμε επιτέλους να έχουμε ανταγωνιστική γεωργία σε όλα τα κράτη-μέλη με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις άμεσες ενισχύσεις μεταξύ των κρατών μελών. Και οι αγρότες στην πατρίδα μου πολύ δύσκολα θα ανταγωνιστούν αγρότες σε άλλα κρατημέλη που λαμβάνουν παχυλότερες άμεσες ενισχύσεις. Η κυρία Εράς Γκαρσία. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους καλεσμένους μας που μας παρουσίασαν τη μελέτη τους. Και Όντως ε, υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο στην ανακοίνωση. Γίνεται λόγος για μια ανθεκτική γεωργία. Το, ο ορισμός του ε, λεξικού για το ανθεκτικός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αντα, ανταπεξέλθει και να ξεπεράσει ε, αντίξουες και τραυματικές συνθήκες. Ενώ εμείς μιλούμε για την ανθεκτικότητα της γεωργίας με θετικό πνεύμα. Ενώ ο ορισμός του που δημιουργεί την αίσθηση ότι μιλάμε για μια κρίση, για κάτι πολύ αρνητικό. Τελικά τι θέλουμε. Ε, αν δεν θέλουμε να πλήξουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, θα, δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε μια αμυγός κοινοτική πολιτική που είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Οπότε από αυτή την άποψη, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να συμφιλιώσουμε μια καλή γεωργική και ισχυρή γεωργική πολιτική, κοινή γεωργική πολιτική, με όλα αυτά τα σχέδια περί επικουρικότητας που μας εξηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συμπεριλάβατε και στη μελέτη σας. Πώς είναι δυνατόν με κάποια σχέδια που μπορεί να είναι περιφερειακά ή εθνικά να επιδιώκουμε έναν ευρωπαϊκό αντικτύπο, ενώ ταυτόχρονα εμ, υποσκάπτουμε το ευρωπαϊκό πνεύμα αυτής της πολιτικής. Πώ είναι δυνατόν να θέλουμε μια ισχυρή κοινή γεωρική πολιτική όταν ο πρόεδρος Γκούγκερ περιλαμβάνει, ε, προτείνει περικοπή 15% στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, στην αγροτική ανάπτυξη. Και η μόνη απάντηση που μας δίνει είναι περισσότερη χρηματοδότηση. Πώ είναι δυνατόν να έχουμε χρηματοδότηση όταν είναι διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες των κρατών μελών για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Πώς πιστεύετε ότι μια τέτοια αντιμετώπιση θα μας ενισχύσει. Το αντίθετο θα μας αποδυναμώσει αυτή η επικουρικότητα και ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόμο για την εξάλληψη της κοινή γεωργικής πολιτικής. Συμφωνείτε? Κυρία Ρας Γκαρσία λέμε ότι η ισχύ της Ευρωπαϊκή Ένωση έγκυται στην πολυμορφία τη, στη διαφορετικότητά της. Γιατί λοιπόν να μην στηρίξουμε την ισχύ τη Ευρωπαϊκή Γεωργίας στην πολυμορφία της γεωργία. Στην ε, πατρίδα σας που έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ε, είναι πολύ ωραία η Γεωργία και έχει λαμπρά αποτελέσματα. αλλά και άλλο είδους γεωργία σε άλλη χώρα, σε άλλη περιφέρεια έχει τα δικά της πλονεκτήματα. Δεν χρειάζεται να έχουμε ομογενοποίηση και απόλυτο ομοιομορφοποίηση. Να επιτρέψουμε την επικουρικότητα, υπό τον όρο βέβαια ότι η επικουρικότητα αυτή δεν θα στρεβλώσει την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ κύριος Μπόκοβιτς. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση και εγώ ε, δεν άκουσα να γίνει κανένα σχόλιο για το κατά πόσο είναι σωστός ο προσανατολισμός της κοινή γεωρικής ε, πολιτικής. Έχω τρεις ερωτήσεις να υποβάλω. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά το πρασίνισμα. Δεν υπάρχει άραγε ο φόβος ότι τελικά αυτό το οποίο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας που λέει ότι τα κράτη-μέλη τα ίδια αποφασίζουν ποια μέτρα θα εφαρμόσουν και ποια όχι. Και αν τελικά ε, προχωρήσουμε προς αυτήν την εξέλιξη ενδέχεται να σκεφτεί μεγαλύτερη πίεση προς την ε, γεωργία. Και η Κομισιόν ε, θα παίξει το ρόλο του πόντιου πιλάτου, δεν θα ανακατευτεί καθόλου. Εγώ όμως ε, διερωτώ με μήπως όλα αυτά τελικά αποτελούν παγίδα για τη Γεωργία. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημά μου. Το δεύτερο, όσον αφορά τους ε, νέους γεωργούς. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε το 2017 πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε συνδυασμό με αυτά που αποφασίστηκαν στην, στον κανονισμό Omnibus ε, που προβλέπει μεγαλύτερες ενισχύσεις για τους ε, νέους γεωργούς. Και ε, σας ερωτώ κατά πόσον θεωρείτε ότι η επαναφορά της σύνταξη στο γεωργικό τομέα ενδεχομένως να οδηγήσει στο να ασχοληθούν περισσότεροι στο μέλλον με τη γεωργία. Τρίτη ερώτηση. εφή χωριά οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες ε, στον τομέα της υγείας και σε άλλους. Ε, ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι τελικά αν προάγουμε την ψηφιοποίηση ενδέχεται να παραμείνει σε καθυστέρηση ο γεωργικός τομέας. Κοιτάξτε, είναι σαν να είμαστε εδώ μπροστά στη γυάλινη σφαίρα και να θέλουμε να ερμηνεύσουμε τι ακριβώ εννοούσε η Κομισιόν με αυτή την περίφημη ανακοίνηση. Αυτό που είναι σαφέ είναι ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλου του στόχου. Δηλαδή και μεγαλύτερη ευελιξία και αύξηση τη παραγωγικότητα και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντο ε, και τήρηση των στόχων της χιλιετίας και προσανατολισμό στην αγορά. Μα δεν γίνεται, δεν μπορούμε να τα επιδιώξουμε όλα αυτά μαζί. Πρέπει να κάνουμε επιλογές. Και εφόσον έχουμε υπογράψει την ε, Συμφωνία για το Περιβάλλον στο Παρίσι, ε, και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα τους επιτύχουμε τους στόχους αυτής της συμφωνίας. Λένε πολλοί να το κάνουν τα κράτη-μέλη προοριτικά, το καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και διαρωτώ με, μα είναι σοβαρό, ε, και πώς θα το κάνουν αυτά τα κράτη-μέλη και πώς θα μετρηθούν οι στόχοι. Για μένα αυτό που παίζει ρόλο είναι να υποβάλλονται προτάσεις. Και λένε οι Βρυξέλλες κάνουν προγράμματα. Και αν ε, δεν εφαρμόζουν τα προγράμματα, ε, τι γίνεται, ποιος τιμωρείται, ο μεμονωμένος Γιώργος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια απόλυτη φούσκα όταν λέμε ότι ναι εφαρμόζονται προγράμματα και αν δεν εφαρμόζονται κανείς δεν τιμωρείται. Δεύτερος πυλώνας, διαχείριση κινδύνων. Εκεί πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Αυτή η περικοπή κατά 25% είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Και ρωτώ, εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα καλό εργαλείο. Μα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχε. Και τελικά το πώς μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά και με λιγότερα κονδύλια, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Κοιτάξτε, λάβαμε μια σημαντική απόφαση. Είδαμε λοιπόν, βασιστήκαμε στην πρόταση της ε, Κομισιόν. Εδώ πέρα όμως το PowerPoint βλέπουμε κάτι το οποίο είναι σχεδόν ανήθικο γιατί ακούγεται πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έχουμε τους στόχους, θα τα εφαρμόσουν τα κρατημέλη. Η Κομισιόν έρχεται σε επαφή μόνο με τα κρατημέλη, ποτέ με τους αγρότες. Κανείς δεν θα ε, πάει πλέον στα χωράφια. Όμως έχω κάποιες ερωτήσεις. Το πρώτο σημαντικό ερώτημα είναι πού βρίσκεται ο αγρότης σε αυτό το σύστημα. Για τον αγρότη κάνουμε πολιτική, μιλάμε για γραφειοκρατία και μείωσή της και αυτή θα πρέπει, βλέπουμε ότι θα γίνει μεταξύ Κομισιών και κράτους μέλους. Πού βρίσκεται ο αγρότης. Δεύτερον, είπατε πως ε, η υπόθεση πάσχει εφαρμογή γιατί εφαρμόζουν τις πολιτικές διαφορετικά τα κρατημέλη και έχουν 27 διαφορετικές απαντήσεις στο κάθε θέμα και μετά ξανά χάρηκα εκεί που είπατε ότι θα έχουμε και αύξηση της παραγωγικότητας καλό οπωσδήποτε αυτό αλλά το ερώτημα είναι τι εννοείται εδώ θα πάνε οι άμεσες πληρωμές προς την αύξηση της ε, παραγωγικότητας αλλά τι θα γίνει μετά με με τις ε, πιο παραγωγικέ επιχειρήσει. Ο κύριο Κολομπιά, έχω μία ερώτηση προ του συντάκτε μελέτη. μελέτης. Πρόκειται για ένα θεμελιώδε ερώτημα που απασχολεί την ε, περιοχή της Νουβέλα Κιτέν, που είναι η πιο ε, ε γεωργική περιοχή της Γαλλίας, που παράγει γνωστά βοηδή, πολύ, πολύ γνωστή φυλή βοηδών, καλαμπόκι και άλλα ε, προϊόντα. Θεωρείτε ότι η νέα πρόταση είναι αποτελεσματική για την ε, γεωργική πολιτική και για την κατάσταση των αγρατών. Και κυρίως είναι αποτελεσματική απέναντι στη γεωργική πολιτική των ε, ανταγωνιστών μας όπως είναι ο γεωργικός νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι κρατικές ενισχύσεις που δίνει η Βραζιλία για παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριος Ρεμπέγκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες σε πάρα πολλά θέματα. Το πιο σημαντικό και ανησυχητικό είναι ότι κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ερήμην των παραγωγών, ερήμην των αγροτών, με το πρόσχημα ότι θα βελτιώσει την κατάσταση στη Γεωργία, ε, διαπιστώνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο. Ε, ούτε τα δικά μα σχόλια λαμβάνει υπόψη στην Επιτροπή, παρόλο που εμεί εκπροσωπούμε το συμφέρον των αγροτών. Ζητάτε περισσότερο συντονισμό. Τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Κάθε φορά που μιλούμε για συντονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να το ερμηνεύει ως ε, ανάγκη επιβολής προγραμμάτων. Κάθε φορά που μιλούμε για συντονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται τι διαφορέ υπάρχουν στη γεωργία μεταξύ των κρατών μελών και τι διαφορέ υπάρχουν μεταξύ των αγροτών των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ανταγωνιστικότητα στο μέτρο που επιτρέπουμε ε, που υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ στι άμεσε ενισχύσει, για παράδειγμα. Πώ θα έχουμε ανταγωνιστικότητα όταν ε, είναι διαφορετικέ οι ενισχύσει οι επιδοτήσεις που δίνονται στα κράτη-μέλη ή είναι διαφορετικό το ύψο των άμεσων ενισχύσεων. Και μιλούμε για ιστορικά δικαιώματα ή για μεταβίβαση, κληρονομική διαδοχή στη γεωργική εκμετάλλευση. Μα αν δεν προσφέρουμε λύση στους νέους γεωργούς, πώς να θέλουν να κληρονομήσουν τη γεωργική εκμετάλλευση και να ασχοληθούν με τη γεωργία. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού είπατε ότι θα χρησιμοποιηθούν ε, μέσα μείωσης ε, του κινδύνου και το λέτε για καλό αυτό. Στις ΙΠΑ είχαν την εμπειρία και φεύγουν από αυτήν την εμπειρία και δεν σημαίνει αυτό αναπόφευκτα λιγότερα λεφτά στην τσέπη του αγρότη. Να σας πω και το εξής. Τελείωσε ένα τουρνουά γκολφ στις ΙΠΑ με βραβείο 5 ή 6 εκατομμύρια δολάρια και δεν τα πήρε κανένας αγρότης. Ο Τάγκερ τα πήρε και όλοι οι άλλοι γκολφέρ. Εδώ πώς θα δουλέψει δηλαδή το σύστημα. Τα λεφτά που πηγαίνουν ε, τώρα στους αγρότες, Πώ πώς θα τα φάνε και εδώ τίποτα τέτοιες εταιρείε. Και κάτι άλλο, μπερδεύουμε το ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα με την αιτιώδη σχέση. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο βεβαίω. Ακριβώς το πρόβλημα είναι ότι προτιμήσαμε κανόνια αντί για βούτυρο. Έχει φάει κανείς σας σφαίρα. Δεν τρώγονται οι σφαίρες. Χόιμπουχ. Κυρία Χόιμπουχ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτερ Γιάρ έθεσε το ερώτημα πού είναι σε όλα αυτά ο αγρότης. Και εγώ το ίδιο λέω, χάνουμε κάθε μέρα δεκάδες αγροκτήματα και εκμεταλλεύσεις. Ειδικά μικρές και μεσαίες. Αν μιλάμε λοιπόν για ανθεκτικότητα σε όλα τα επίπεδα, οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό, τότε χρειαζόμαστε καλές γεωργικές δομές για τους μικρομεσαίους αγρότες. Υπάρχει μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Γητίνγκης ε, η οποία είδε ακριβώς το θέμα της βιοπικιλότητας και μία μικρή αγροτική εκμετάλλευση έχει πολύ περισσότερη βιοπικιλότητα ενώ σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις χάνεται η βιοπικιλότητα και τώρα πλέον αυτό αποδεικνύεται. Γιατί λοιπόν στην ανάλυση σας δεν εμφανίζεται καθόλου η δομή των εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ. Κυρία Σλάιρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ το ερώτημα του Πέτερ Γιάρ να κάνω, αλλά έχω και άλλη μια ερώτηση ε, μετά από αυτό το οποίο έκανε η Έστερ Χέρανς ε, Εγώ συμφωνώ εδώ πέρα μαζί σας, αλλά μην ξεχνάτε και το εξής. Οι πολυεθνικές που συνεργάζονται με τους αγρότες θα δούνε που πάνε οι επιδοτήσεις και εκεί ακριβώς θα κατευθυνθούν και αυτή ακριβώς είναι και η ευριανή μου τροπολογία. Να δούμε δηλαδή ακριβώς πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλες και σοβαρές ανησυχίες. Να δούμε επίσης πώς έχουν οι επιδοτήσεις στις διάφορες ε, χώρες ε, και ποιο είναι το κόστος ε, των αγροτών. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις ε, πριν, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να κάνω εγώ κάποιες σκέψεις. Ε, καταρχήν να δούμε αν τα κονδύλια της γεωρικής, ε, του γεωρικού προϋπολογισμού αξιοποιήθηκαν καλύτερα. Έπιασαν τόπο, έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων για να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και να πιάνουν περισσότερο ε, τόπο οι επενδύσει. Αλλά αυτό θέλουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή μήπω θέλουμε ε, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα με συγκέντρωση ή χωρίς. Οπότε θα πρέπει να διατηρήσουμε το γεωργικό μοντέλο μας. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη. Αν έχουμε συγκέντρωση θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί το γεωρικό εισόδημα. Εμείς όμως ταυτόχρονα θέλουμε να διαφυλάξουμε το γεωργικό μας μοντέλο εξασφαλίζοντας τα γεωργικά εισοδήματα. Τι ακριβώς ε, είναι, ποιος ακριβώς είναι ο στόχος μας, τι ακριβώς είναι το ζητούμενο εδώ. Επίσης, τι εργαλεία χρειαζόμαστε. Γιατί όταν καθορίζουμε τους στόχους, τις αρμοδιότητες, τις λειτουργίες. Πώς θα εξασφαλίσουμε τον κοινό χαρακτήρα της κοινή γεωργικής πολιτικής όταν έχουμε τόση μεγάλη ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και από άποψη κλιματική και από άποψη φυσικών ε, συνθήκων και από άποψη παραδόσεων. Τελικά αυτή η διαφορετικότητα, αυτή η ποικιλομορφία είναι προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ή πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι ε, πλεονέκτημα, αξία. Οπότε θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό είμαι υπέρ της ελαστικότητας και είμαι υπέρ της επικουρικότητας. Γιατί λέμε δεν έχουμε στόχους ε, και αρμοδιότητες στα πλαίσια του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί θα προτιμούσαμε με κάθε λεπτομέρεια η ευρωπαϊκή πολιτική να μας ε, καθορίζει τους στόχους ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής, τότε δεν θα έχουμε ε, αυτόνομη δραστηριότητα. Θα, μας, θα επηρεάζει την οικονομική ελευθερία αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια προσδιορίζει τους στόχους και τις μεθόδους υλοποίησης των στόχων. Οπότε ε, καλό είναι να είμαστε και λίγο λογικοί και να δείξουμε κατανόηση. Επίσης, ε, επιδοτήσεις για τους νέους αγρότες. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε κάποια θεμέλια στην οικονομία. Ποιος θα εγγυηθεί την αγορά αγροτεμαχίων, α, κτίριων, γεωργικών μηχανημάτων θα προβλέψουμε κάποια κονδύλια για τη στήριξη των νέων. Αλλά εδώ μιλούμε τώρα για άλλη κλίμακα παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστεί ένας νέος ιδιοκτήτης ε, που θα δημιουργήσει μια παραδοσιακή ε, εκμετάλλευση, αλλά θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα κονδύλια. Επίσης, Μιλούμε για τις νέες προκλήσεις, για την ανάγκη περικοπής του γεωργικού προϋπολογισμού λόγω του χρηματοδοτικού κοινού των Brexit. Το καταλαβαίνω. Αλλά τι γίνεται με τη γεωργία μας. Υπάρχει ένα επίπεδο γεωργικού εισοδήματος που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των γεωργών. Μπορούμε να επιτρέψουμε μείωση του γεωργικού προϋπολογισμού δεδομένης αυτής της κατάστασης. Τι θα γίνει με τη γεωργία μας αν οι αγρότες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Επίσης έχουμε τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργία και που δεν είναι και πολύ ευνοϊκή αυτή τη στιγμή για τους Γιώργους. Είδαμε την περίπτωση της Βραζιλίας. Εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας προβληματιζόμαστε με όλα αυτά τα θέματα. Γιατί δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει κατανόηση για την ε, κοινή ε, γεωργική πολιτική. Ε, αρχίζουν και ασχολούνται με την, Ευρω... με την γεωρική πολιτική στο Κοινοβούλιο μόνο όταν ανακύπτουν κάποια προβλήματα, όταν ανακύπτει κάποια κρίση, όταν έχουμε έλλειψη κάποιων τροφίμων. Τότε θυμούνται όλοι και στο Κοινοβούλιο ακόμη την Επιτροπή Γεωργίας. Ενώ μερικοί λένε τι χρειάζεται τη γεωργία. Μα τη χρειαζόμαστε για να έχουμε επιστηστική ασφάλεια και υγιεινά τρόφιμα. Μου δίνει ένα χαρτάκι ο γραμματέας και μου λέει ότι πρέπει να βάλω τελεία και να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, με ανησυχείτε. Εγώ θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές για τη μελέτη τους. Ε, ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας έδωσε αυτήν την επισκόπηση ε, για την ανακοίνωση. Λοιπόν, τρία σχόλια. Καταρχήν όσον αφορά τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και μετά το περιεχόμενο της έκθεσης. νομίζω ότι εμείς όταν ε, εξετάσαμε την ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε στις 29 Νοεμβρίου, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να μην την ε, αποκόψουμε από διάφορα άλλα έγγραφα με αναλύσεις ε, ότι θα έπρεπε και αυτή η ανακοίνωση να ενταχθεί στις διάφορες αναλύσεις. Και έτσι μετά από κάποιες εβδομάδες δημοσιεύσαμε την αξιολόγηση για τα μέτρα πρασινίσματος, σημαντικό αυτό, και η Παγκόσμια Τράπεζα κατέθεσε μια σημαντική μελέτη για την απόδοση της ε, γεωργικής πολιτικής και για την κατάσταση στις αγροτικές περιοχές. Όταν λοιπόν εξετάσαμε αυτή την ανακοίνωση, όπως επίσης ε, και τις αναλύσεις ε, ε, που σχετίζονται, ας μην ξεχνάμε ότι αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η διαδικασία συνεχίζεται. Μετά από κάποιες εβδομάδες θα καταθέσουμε νομοθετικές προτάσεις και μαζί με τις προτάσεις θα καταθέσουμε και τη μελέτη αντικτύπου που θα συνοδεύουν τις προτάσεις με πολλά στοιχεία που είμαστε σίγουροι ότι θα εμπλουτίσουν τη συζήτηση και θα προσφέρουν τροφή για σκέψη. Παρεπιπτόντως, η μελέτη αντικτύπου θα περιλαμβάνει πολλά παραρτήματα, μεταξύ αυτών ένα παράρτημα που θα περιλαμβάνει ε, τις δημόσιες διαβουλεύσεις, ε, τις απόψεις διαφόρων ε, θεσμών. Μιλάμε τώρα για μία ανακοίνωση του Νοεμβρίου, ενώ το μεταξύ έχουν προκύψει πάρα πολλά. Και πιστεύουμε ότι θα είχε νόημα όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη σας για να γίνει πιο σταθερή η ανάλυση, πιο εμπεριστατωμένη. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Όταν θα έχουμε την έκθεση θα την αναλύσουμε λεπτομερώς. Πρέπει να περιμένουμε κάποιες εβδομάδες για να έχουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής. Και το λέω αυτό γιατί σας λέω, εδώ πρόκειται για ανακοίνωση, δεν πρόκειται για ε, πρόταση. Πολλοί άκουσα, ε, μιλάνε για ε, πρόταση της Επιτροπής. Δεν είναι έτσι, πρόκειται για ανακοίνωση, για να περιχαρακωθεί η συζήτηση, αλλά οι νομοθετικές προτάσεις θα κατεθούν μετά από κάποιε εβδομάδες, όπου θα ληφθούν υπόψη διάφορες απόψει και αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκφράστηκαν τους τελευταίους μήνες. Όσον αφορά τώρα την ανάλυση των κυρίων καθηγητών, δεν τις αμφισβητούμε, τις αναλύσεις, κυρίως εκεί που τοποθετούνται ε, σχετικά με τις ε, προκλήσεις που προκύπτουν. Θέλω όμως να υπογραμμίσω τρία θέματα όπου διαφωνούμε. Το πρώτο αφορά στην κριτική που ασκήσατε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ε, άμεσες ε, πληρωμές. Εμείς πιστεύουμε ότι η άποψη που εκφράζεται εδώ είναι λίγο περιοριστική με, σχετικά με τον τρόπο που παίζουν αυτές οι άμεσες ενισχύσεις. Ε, ε, δηλαδή αυτές ε, δεν είναι μόνο για να βελτιώνουν το εισόδημα, αλλά για να υπάρχει και κάποια προστασία για το περιβάλλον. Αυτή η αλληλένδεση του οικονομικού και του περιβαλλοντικού στοιχείου στις ε, πληρωμές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γιατί αν βλέπουμε τις ε, πληρωμές μόνο κάτω από οικονομικό ε, πρίσμα για το αν ενισχύουν το εισόδημα, τι γίνεται με την παραγωγικότητα, αν το κάνουμε αυτό τότε χάνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης εικόνας. Και αυτά σχετίζονται πάλι και με το ρόλο του πρασινίσματος και με το ρόλο του ε, αρχιτεκτονήματος. Εμείς στην Κομισιόν είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να διατηρηθούν οι άμεσες ενισχύσεις, όχι μόνο για να βελτιώνεται το εισόδημα και να υπάρχει σταθερό εισόδημα για τους γεωργούς, αλλά και για να προσφέρεται περιβαλλοντική προστασία. Και κάτι άλλο. Ε, κατά τη, στην έκθεση και μετά στη συζήτηση έγινε επανειλημμένα λόγος για τους νέους γεωργούς, που προφανώς και είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι στη δική μας την ανακοίνωση, αλλά και ε, στις δικές σας τις ε, παρεμβάσεις και τις προφορικές ε, και με τις εκθέσεις που καταθέσατε, οι νέοι γεωργοί αντιμετωπίζονται και στους δύο πυλώνες και νομίζω ότι και οι δύο πυλώνες που πρέπει να συμβάλλουν στην ανανέωση των γενναίων. Η ανακοίνωση δεν αναφέρεται μόνο στον ένα πυλώνα, τον αντίον αναφέρεται και στους δύο πυλώνες και στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους ε, δύο πυλώνες και βεβαίως και στις δράσεις των ε, κρατών μελών. Και ένα τελευταίο σχόλιο που αφορά στο θέμα των ε, ίσων ευκαιριών. Έγινε πρώτα λόγο στη συζήτηση και μετά στην έκθεση. Το μοντέλο που έχει σκεφτεί η Επιτροπή είναι το εξής. Θα υπάρχουν απαραίτητες διασφαλίσεις για να διαφυλάσσονται οι ίσες ευκαιρίες για όλους. Και κάτι που είναι και σημαντικό για την συζήτηση. Κάποιος Κάποιος αναφέρθηκε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αυτό αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τους κανονισμούς. Η Κομισιόν δεν είναι εκείνη που εγκρίνει τις αποφάσεις των κρατών μελών για τις ε, συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αυτές στο μέλλον θα εντάσσονται στο στρατηγικό όμως πλαίσιο της Επιτροπής, άρα δηλαδή τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίζει κάποιο ρόλο όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες ε, περιβαλλοντικές ε, προϋποθέσεις. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν κάποιες εξαιρέσεις και να τις ανακοινώνουν στην Επιτροπή, αλλά δεν είναι εκείνη η Επιτροπή που ε, απαγορεύει ή αποφασίζει. Στο μέλλον όμως όλα αυτά ε, θα εντάσσονται στο στρατηγικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή αν θέλετε στο μέλλον εμείς θα παίζουμε περισσότερο ρόλο και θα ελέγχουμε το τι θα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Ήθελα απλά να τα προβάλλω αυτά τα στοιχεία για να διευκρινίσω την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ανοιχτοί ως προς τη συζήτηση. Όταν η έκθεση θα λάβει την τελική της μορφή, με μεγάλη μας χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις με τους καθηγητές και θέλω να επιμείνω στην ε, δημοσίευση των νομοθετικών προτάσεων. Πιστεύω ότι η έκθεσή μας που θα δημοσιευθεί θα περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία, αναλυτικά και άλλα, που θα είναι χρήσιμα και για το από ακαδημαϊκή σκοπιά, αλλά και από πλευρά, ε, πλευράς χάραξης πολιτικής. Σας ευχαριστώ, γιατί πολύ εύστοχα προσεγγίσατε το πρόβλημα. Για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει περισσότερο λόγο στην εξέταση των στρατηγικών εθνικών σχεδίων. Γιατί αν μια χώρα δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα κονδύλια για να υλοποιήσει ε, το στρατηγικό της σχέδιο, φυσικά θα χρειαστεί μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό θα είναι λοιπόν και αυτά τα στοιχεία να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια ουσιαστικά στοιχεία. Και τέτοιες περιπτώσεις θα έχουμε. Και όλα αυτά θα τα βρούμε και μπροστά μας σίγουρα. Και τώρα ο λόγος καλεσμένους μας. Πέντε λεπτό καθένας παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, Έχετε το λόγο ποιος από τους δύο θέλει πρώτος να μιλήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαρά άκουσα την συζήτηση αυτή. Να ξεκινήσω με αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν. Πράγματι, η Κομισιόν βασίζεται σε ε, αρκετά καλά στοιχεία. Βοήθησα και εγώ να γράψουμε την αξιολόγηση των μέτρων πρασινίσματος. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να χαράζουμε πολιτική με βάση τα στοιχεία και είναι δύσκολο. Για τις άμεσες πληρωμές, ναι, κατάλαβα τι λέτε, αλλά αν δεχτούμε ότι τα λεφτά των άμεσων πληρωμών αγοράζουν κάτι για το περιβάλλον, για την νέα αρισιμότητα, πρέπει να μπορούμε να την δούμε αυτή την αρισιμότητα και να σχηματίσουμε άποψη για την ποιότητά της. Είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο αν δεν την ξέρουμε την λεπτομέρεια αυτής της πολιτικής, οπότε για την ώρα θα μου επιτρέψετε να είμαι κάπως επιφυλακτικός. για τους ίσορους ανταγωνισμού. Το είπε και ο κύριος Ντόρφμαν. Σε ποιο βαθμό θα υπάρχει η δυνατότητα να αποκλίνουν αυτά τα σχέδια στο τι προτείνουν, στο ποιες προτεραιότητες έχουν κτλ. Και πάλι λοιπόν με τα λίγα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Εάν οι στόχοι όπως ίσως το περιβάλλον υποβαθμιστούν ή ίσως υποβαθμιστούν στο πλαίσιο των δύσκολων πολιτικών της στήριξης του εισοδήματος ε, των αγροτών, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει περιθώριο μιας περιχαράκωσης των κονδυλίων, όπως είχε γίνει με τα πράσινα μέτρα στην τρέχουσα γεωργική πολιτική. αυτά τα οποία είπαμε για την ένταση μεταξύ περιβάλλοντικών μέτρων και εισοδήματο των αγροτών. Μπορεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούν να ληφθούν περιβαλλοντικά μέτρα που βελτιώνουν το εισόδημα. Τα ψυχανθή, παραδείγματο χάρη, τα οποία βεβαίω έχουν και συνδεδεμένη στήριξη, αλλά βεβαίω χρησιμεύουν και ως ε, μεταλλικά λιπάσματα για άλλες καλλιέργειες. Οπότε τα πρωτεϊνούχα και τα ψυχανθή είναι κάτι το οποίο είναι αμοιβαία επαφελές και για το περιβάλλον και για τους αγρότες. Βεβαίω ε, πάντα σύμφωνα με τις ε, σχετικές μελέτες. Άλλη ερώτηση που έγινε, αν υπάρχει εδώ πέρα δηλαδή κάποια μεταρρύθμιση. Ναι, αλλά θα είναι αρκετά δύσκολη, απαιτεί φαντασία και αλλαγή επίσης ε, των σχετικών ε, νοοτροπιών. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες ε, γίνονται πιο επιδέξεις στην χρήση τεχνολογίας, γνώσεων και έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν οι σχετικέ αποφάσει για να είναι βιώσιμε και οι καλλιέργειε. Αναφέρθηκαν οι περιφερειέ, ναι, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν αυτά τα στρατηγικά σχέδια εκεί όπου υπάρχουν περιφερειές. Τα ομοσπονδιακά κράτη-μέλη προφανώς έχουν διάκριση εξουσιών, οπότε στην Γερμανία το ομοσπονδιακό κράτο είναι υπεύθυνο για τον πυλώνα 1 και τα κρατήδια για τον πυλώνα 2 και θα είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα επί της αρχής μπορεί να γίνει, αλλά σημαίνει ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο και εμπιστοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να εξασκηθούμε αρκετά. Αυτά ήθελα εγώ να πω. Θα δώσω τον λόγο στον Κριστόφ για να πει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην έκθεση αυτή λοιπόν που θα λάβετε προσπαθήσαμε να μείνουμε καθαρά τεχνικοί και να μην δώσουμε μία προσωπική ε, άποψη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ζητήματα για τα οποία μας ζητήσατε άποψη, οπότε μπορώ να γίνω πιο υποκειμενικός προφορικά. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις που έλεγαν αν υπάρχει πραγματικό όραμα της Κομισιόν, αν υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής επικουρικότητας και μίας κάπ λιγότερο κοινή. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος και συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Ντεκάστρο. Και βεβαίω πρέπει να τα δούμε αυτά ανάλογα με την αφετηρία θυμάμαι ήμουν στο Συμβούλιο της Νανσί όπου υπήρχε ε, ένα κοινό όραμα για την Γεωργία, αλλά αυτό πλέον δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνε της. Γεγονός είναι πως ε, χοντρικά στέλνει όλα τα προβλήματα στα κράτη-μέλη, δηλαδή οτιδήποτε είναι δύσκολο, οτιδήποτε κοστίζει, το ξεφορτώνεται. Αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος νομίζω για το μέλλον, ειδικά αν δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα είναι αρκετά αυστηρό ή κοινό όσον αφορά τα δημόσια αγαθά όπως το περιβάλλον. Για να πάμε στην ε, πρόταση της ε, Κομισιόν. Αλλά ίσως ε, έτσι να θέλει μια πιο συντηρητική κυβέρνηση, μια χώρα να πάει στις επενδύσεις, μια άλλη κυβέρνηση αλλού, στις συνδεδεμένες πληρωμές, μια τρίτη κυβέρνηση κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η ε, δυνατότητα και να σκεφτούμε τελικά ε, αξίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνει μια πολιτική η οποία δεν θα έχει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτά για το θέμα αυτό, για την παραγωγικότητα και την σύγκρουση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ μιας πιο βιώσιμης και μιας πιο παραγωγικής γεωργίας. Δεν είναι οπωσδήποτε αντιφατικό αυτό βεβαίως γιατί η παραγωγικότητα μετριέται και με το ποιοι είναι οι παραγωγικοί συντελεστές που μπαίνουν, αν θέλετε, για την παραγωγή και μπορούμε να έχουμε μια γεωργία, όπως λέμε, στα γαλλικά τα ωραία έτσι πιο αυτόνομη και με μεγαλύτερη οικονομία μέσων. Κάτι το οποίο βεβαίως θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ένα τέτοιο κοινό πλαίσιο για να ενθαρρυνθεί αυτή η κατεύθυνση στην μελλοντική ΚΑΠ. Για αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Μαγκίνες για την σημασία των άμεσων πληρωμών και τον κίνδυνο μείωσής τους, πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου πως αυτή η εξάρτηση του εισοδήματος από τις άμεσες ε, πληρωμές ε, έχει δημιουργηθεί εν μέρει από τους ίδιους αγρότες. Να αφαιρθώ σε μια περιοχή την οποία γνωρίζω καλά που οδηγήθηκε στην ορεινή κτηνοτροφία λόγω των ενισχύσεων του γαλλικού κράτους με πολύ ε, με εδάφη πολύ και χώματα πολύ ψηλά, καθόλου βαθιά, καθόλου αζωτούχα και τώρα ε, βλέπουμε ότι έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή να λαμβάνουν 6-10 ευρώ το εκτάριο και πραγματικά τσέτερης πάρυμπους, εάν υπάρξει μείωση των αμέσων πληρωμών, θα υπάρξει και μία μείωση κάποιων καλλιεργούμενων εδαφών. Τώρα, για την αναγκαιότητα του να υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο πολύ πιο κοινό, εδώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο οδηγεί σε έναν ε, κίνδυνο να μην πάμε τελικά στο πρασίνισμα, ειδικά αν μιλάμε για το πρασίνισμα στο σύνολο των ε, πληρωμών ε, μετά τη μεταρρύθμιση του 2013. Ακόμα και αν περιμένουμε να δούμε βέβαια ποια θα είναι η αιρεσιμότητα του πρώτου πυλώνα στην πρόταση της Κομισιόν, υπάρχει ένας κίνδυνος οπισθοδρόμησης στο μέτωπο αυτό. Ευχαριστώ. Ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο προς τα πίσω. Το θέλουμε. Επίσης, οι περισσότεροι θα θέλουν να χρηματοδοτήσουν τη γεωργική πολιτική. Ναι, αλλά αν λάβουμε υπόψη τι χρηματοδοτείται με την κοινή γεωργική πολιτική, διαπιστώνουμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη και την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας. Γιατί μιλούμε για τέτοιες διαστάσεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ολοκληρωμένη μελέτη. Και σίγουρα υπό την ε, επιρροή ο συντάκτης γνωμοδότης Επιτροπής Γεωργίας είναι ο κύριος Ραμόν Λουίς Βαλκάρσελ Σίσο, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή γενικό προϋπολογισμό του 2019. Διότι από τους σοσιαλιστές και ρουμπίχα από το ΕΛΚ. Και μάλιστα όσοι ήθιστε και θα σας δώσουμε σε λίγο το λόγο αφού ακούσουμε και τον συντάκτη της γνωμοδότησή μας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι κύριε Βιώτη. Κύριε Σίσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντανιέλ Βιώτη που έχει την καλοσύνη να έρθει στην Επιτροπή μας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που είναι αναφυσβήτητα πολύ σημαντικό. Οι αγρότες επλήγησαν τα τελευταία χρόνια. Ε, φοβερή αστάθεια και των τιμών ε, απαναφισβήτητα πολύ σημαντικό. Οι αγρότες επλήγησαν τα τελευταία χρόνια. Ε, φοβερή αστάθεια και διακύμα των τιμών, ε, απάτες ε, και καταχρήσεις που έγινε στην αλυσίδα τροφίμων, φτώχυνση του αγροτικού πληθυσμού. Είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 2019. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανησυχίες και προβληματισμό για το ε, τι ε, ε, συνέπεια θα έχει οποιαδήποτε, κάποια αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα επηρεάσει μετά από πολλά χρόνια εξαιρετικών διακοιμάσεων η έλλειψη παράταση των μέτρων ίσως επιδεινώσει την κατάσταση των κλάδων και βράχει και μεσοπρόθεσμα. Επαναλαμβάνω, αν δεν παραταθούν τα μέσα αντιμετώπισης του ρωσικού εμπάργου. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη βράχη και μεσοπρόθεσμα. Επαναλαμβάνω, αν δεν παραταθούν τα μέσα αντιμετώπιση του ρωσικού εμπάργου. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη απόρριψη μου, κατηγορηματική απόρριψη μου ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει 5% περικοπή των κονδυλίων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαφυλάξει το γεωργικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ, γιατί ήδη στο παρελθόν έχει υποστεί πολλές μειώσεις και περικοπές. Πολλά δε μάλλον που επιβάλλουμε πιο απαιτητικές ε, διατάξεις προς τους ευρώτες μας εν ώψη της, ΚΑΠ, της νέας ΚΑΠ. Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε τον γεωργικό πληθυσμό στην Ήπεθρο και να ε, συνεχίσει η γεωργία μας να πληρεί υψηλέ προδιαγραφές ποιότητας και επιστηστικής ασφάλειας, θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρωταρχικό μήνυμα που θα ήθελα να διαβιβάσω στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Σε δευτερολογήσετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρο και την Επιτροπή σας ε, για την ε, φιλοξενία που μου προσφέρουν. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο γιατί πηγαίνω στι διάφορε επιτροπέ. Μετά πρέπει να πάω σε μια άλλη επιτροπή για να παρουσιάσω τον προπολογισμό. Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για αυτό. Δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σας και τον συνάδελφο κ. Ντόρφμαν για την ε, θέσπιση σήμερα το πρωί της έκθεσης πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το στηρίζω και το λέω αυτό απλά για να ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. Ντόρφμαν να ξέρει ότι στηρίζω και εγώ τη δική του τη δουλειά. Ε, από πλευράς μεθόδου θα ήθελα να διευκρινίσω ε, και εδώ αυτό που θα πω και σε άλλες επιτροπές, ότι για μένα σε αυτή τη φάση ακούω. Ακούω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν έχουμε ούτε καν το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν έχουμε ούτε καν το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θα παρουσιαστεί το σχέδιο αυτό στις 23 Μαΐου την επόμενη εβδομάδα. Άρα δηλαδή μιλάμε περισσότερο υποθετικά και όχι πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα. Όμως η δική μου η πρόθεση ε, όσον αφορά στο τόσο σημαντικό ρόλο που έχω αναλάβει ως ε, εισηγητής του Γενικού Προεπλογισμού Η δική μου πρόθεση είναι να επιτύχω τη μέγιστη δυνατή συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Προφανώς και θέλω να με στηρίξουν οι πολιτικές ομάδες, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι το θεσμικό στοιχείο. Δηλαδή να έχω την υποστήριξη όλων των επιτροπών και ως εκ τούτου θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ σε όλα αυτά που θα μου ζητήσουν οι επιτροπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας για αυτά που είπε. Ε, εγώ στις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, που ψηφίσαμε το Μάρτιο ε, προσπάθησα να προβάλλω ότι είναι σημαντικό σε κατευθυντήριες γραμμές που ψηφίσαμε το Μάρτιο προσπάθησα να προβάλλω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική και αυτό όχι μόνο διότι σημαίνει την ε, μια οργών. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω έχει σχέση με τη σημασία της ε, γεωργίας και των γεωργικών πολιτικών ε, σε σχέση με, την, με τον γενικότερο προϋπολογισμό. Πρέπει να στηρίξουμε ένα τομέα που είναι καθοριστική σημασία από οικονομική σκοπιά. Θα υπάρχει άμεση σχέση του προεπλογισμού του 2019 με το Brexit. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε ε, με την Επιτροπή σας για τον προεπλογισμό του 2019 έτσι ώστε να υπάρχουν ευβίωνες προπτήσεις ε, του επόμενου πουδουπού αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να εργαστούμε καλά και αποτελεσματικά για θέματα γεωργίας ε, και περιβάλλοντος σε αυτόν τον ε, προπλογισμό. Αυτό είναι ε, καθοριστική σημασία και για να επαναφέρουμε αυτά τα οποία λόντως ε, σε αυτόν τον προπολογισμό. Αυτό είναι καθοριστική σημασία και για να επαναφέρουμε αυτά τα οποία... Να σας υπενθυμίσω κάποια επίκαιρα θέματα για τον προϋπολογισμό του 2019. Δυστυχώς, εσχύριο κρέατος, ε, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη επαρχία, αλλά και από άλλες επαρχίες της Ουγγαρίας. Οπότε, οι χώρες της Βαλτικής, η Σλοβακία, η Ρουμανία θα επηρεαστούν από το προκαλέσει ε, αυτή η ζωονόσο. Γι' αυτό σα παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Κυρία Τακάινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός για το 2019 είναι πολύ σημαντικός ε, για το γεωργικό τομέα. Τώρα εστιάζουμε την προσοχή μας περισσότερο στο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά ο προεπλογισμός πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον στο ίδιο ύψος όπως και προηγούμενος, διότι η κατάσταση των γεωργών είναι πολύ δύσκολη, ε, οι γεωργοί εισοδηματικά βρίσκονται στο 40% των υπόλοιπων τομέων. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε κυρίως με τις ε, μειονεκτούσες ε, περιοχές και να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στην ευημερία των ζώων και στην ποιότητα των τροφίμων. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον μας, χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και νέους γεωργούς. Θέλω λοιπόν κάτω από το πρίσμα αυτό να προβάλλω το θέμα των αγορών γάλακτος στον προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας προβλήματα ε, εισαγωγής ε, που σχετίζονται με τη Ρωσία. Δεν είναι δυνατόν αυτό να αγνοείται στον προϋπολογισμό η γαλακτοπαραγωγή, κυρίως στη Φινλανδία αλλά και στις άλλες χώρες της Βαλτικής, υποφέρουν από τις χαμηλές τιμές παραγωγής. Παρά τις ε, προσπάθειες ε, ε, δεν μπορέσαμε να αντικαταστήσουμε τη Ρωσία ως χώρα προορισμού των προϊόντων μας. Οι αγορές, πραγματικές αγορές δυστυχώς μείωσαν την τιμή του γάλακτο σε πάρα πολλές χώρες. Ως εκ τούτου θα πρέπει στον προϋπολογισμό να υπάρχει μια τέτοια πρόταση που θα προστατεύει τους παραγωγούς από την υπερθέρμανση των αγορών και από τις σχέσεις με τη Ρουσία και παρεπιπτόντως να ανανεώσουμε και τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων σε αυτό τον τομέα για να μην υπάρξει περίκο πολύ γρήγορα. Ε, πρώτα απ' όλα και εγώ ευχαριστώ ε, το συνάδελφό μας, ε, το Ραμοντουή. Σε ευχαριστώ και τον Ντανιέλ Βιώτη που μας βοηθάει σε αυτή την προσπάθειά μας ως Επιτροπή Γεωργίας για να υπερασπιστούμε τον προεπολογισμό της ΠΑΚ. Ο Ραμόν είπε ότι εμείς σε αυτή την Επιτροπή ε, δεν αντιζητάμε περισσότερα για τους γεωργούς με το πρασίνισμα και με όλα τα άλλα που πρέπει να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν, ε, ζητάμε από τους γεωργούς ε, νέα πράγματα, υποχρεώσεις, όμως υπάρχει πρόβλημα στον προπολογισμό και ε, υπάρχουν περικοπές. Ε, γνωρίζουμε βέβαια ότι κάποιες περικοπές οφείλονται στην έξοδο ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και ερωτώ, ε, και δεν καταλαβαίνω, γιατί οι γεωργοί να πρέπει να πληρώσουν για μια νόμιμη τελικά απόφαση των Βρετανών. Τους επιβάλλουμε περισσότερες υποχρεώσεις, αλλά τι κάνουμε, τους περιορίζουμε τις πληρωμές. Ευχαριστώ. οι συνάδελφοι της ΔΕΒΕ θα πούν δεν θα κάνουμε αυτές τις περικοπές. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την ανταγωνιστικότητα και τη, μάλλον την συνεισφορά των κρατών μελών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αν είχαν αυξηθεί οι εθνικές συνεισφορές κάποιο χώρο μελών δεν θα είχαμε σήμερα προβλήματα. Προσοχή λοιπόν που προτείνουμε προ... περικοπές. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε στην Ρουμανία θέλουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει και στις μεγάλες και στις μικρές γεωρικές εκμεταλλεύσεις να λάβουν των αγροτικών περιοχών. Κάτι που απευχόμαστε. Ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα πρωτότυπο να πω ε, και μάλιστα ο προπολογισμό του 2019 σε σχέση με αυτό που μας ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προπολογισμό μετά το 2020 ε, θα πρέπει να ε, μας εστιάσει περισσότερο στο θέμα της επιστηστικής ασφάλειας και βλέπουμε ότι τεράστιες διακοιμάσεις υπάρχουν στις τιμές και μια κρίση που δυστυχώς δεν καθυσυχάζεται ή δεν αντιμετωπίζεται με τα κονδύλια του προπολογισμού. Και έχουμε και το ρωσικό εμπάργκο που φαίνεται να αγνοείται από τον προϋπολογισμό του 2019. Έχω όμως σοβαρότερες ανησυχίες. Τις ανέφερε και ο κύριος Δεκάστρο. 31 Μαρτίου 2019 δεν έχουμε πια μαζί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε τις συνέπειες αυτής εξόδου στον τομέα του κρέατος, για παράδειγμα θα είναι μεγάλο το διακύβευμα λοιπόν και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ήδη από το 2019 γιατί οι σημερινές κρίσεις ε, είναι πολύ διαφορετικές από τις μελλοντικές Ίσως λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα ψηλότερο προϋπολογισμό το 2019 για να μην έχουμε μια δραματική εξέλιξη για τον γεωργικό πληθυσμό. Και λόγω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που υποθέτω ότι δεν ε, αναμένεται να απαντήσω σε αυτά τώρα. Γιατί αυτά μπορεί να γίνουν ε, αλλού με τρόπο. Λοιπόν, για να είμαι σαφής. Η πρόταση που κάνουμε για τον προπολισμό τα κάνει βασίζεται σε 28 κράτη-μέλη. Κοιτάμε λοιπόν προσεκτικά τις εξελίξεις και βεβαίως εάν υπάρχουν βεβαιότητες για το 2019 η Κομισιόν θα είναι έτοιμη να φέρει έναν διορθωτικό προϋπολογισμό στην χειρότερη των περιπτώσεων. Οπότε αυτή τη στιγμή βασιζόμαστε σε ένα σενάριο 28 χωρών. Εάν όμως συμβεί κάτι είμαστε διατεθειμένοι να καταθέσουμε έναν διορθωτικό προπολογισμό πάντα σε συνεννόηση με σας. Οι άλλες ε, παρατηρήσεις αφορούσαν το ρωσικό εμπάργο. Στην ανάλυση μας εμείς, οι άλλες ε, παρατηρήσεις αφορούσαν το ρωσικό εμπάργο. Στην ανάλυση μας εμείς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το εμπάργο αυτό ε, μην ε, ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και αναζητούμε ε, λύσεις μέχρι να επανέλθουμε στην ομαλότητα. Οπότε ο προπολογισμό του 2019 αυτή τη στιγμή δεν προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για τις συνέπειες του ρωσικού εμπάργου. Όσον αφορά τώρα το τρίτο, στη την στιγμή δεν υπάρχει βάση για κάποια συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και πάλι Εάν υπάρξουν συνέπειες λόγω της αφρικανικής γρήψης χείρων ή σε οποιαδήποτε κατάσταση έχουμε το αποθεματικό κρίσεως ε, που υπάρχει ήδη σήμερα για το 2019. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής ο κύριος Βιώτη θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως υποπτευόμουν και σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό το να συμμετέχει κανείς σε αυτή τη συνεδρίαση γιατί το να ακούσει κανείς τα τεχνικής φύσεως θέματα, τα πολιτικά αλλά και τα πιο συγκεκριμένα του κάθε μονομένου θέματος αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό βεβαίως σημαντικό να είναι κανείς εδώ και είναι και πολύ σημαντικό η Επιτροπή Γεωργίας με ε, άτυπο ή με επίσημο τρόπο να είναι πάντα σε επαφή μαζί μου για να με βοηθήσει να καταλάβω και εγώ τις ε, ιδιαιτερότητες του προϋπολογισμού ε, και τις συγκεκριμένες γραμμές που ήταν η πρώτη και δεν ήταν σίγουρα και η τελευταία από πολιτική σκοπιά θέλω να σας πω ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι οι σχέσεις ε, με τα κράτη-μέλη τον ε, Οκτώβριο-Νοέμβριο όταν θα είμαστε στις ε, συνδιαλλαγές. Εγώ έχω κάνει την εμπειρία τεσσάρων συναπτών συνδιαλλαγών που έγινε λόγος για την περικοπή κονδυλίων. Εγώ θα καλέσω όλους τους συναντέλφου μου, όχι μόνο από την Επιτροπή Υπεροπλογισμών, αλλά και από άλλε επιτροπές, να παρέμβουν στις κυβερνήσει τους ε, για να τι ε, πείσουν ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε. Ευχαριστώ και σύντομο σχόλιο και από το συντάκτη γνωμοδότηση από κλιματικές συνθήκες, θεομηνίες, ανοβρία. Και από αυτή την άποψη μας μίλησε ε, για την προσπάθεια περιορισμού των αρνητικών συνεπειών του ρωσικού εμπάργου. Αλλά έχουμε και άλλες δυσκολίες που προκύπτουν από αντίξωες καιρικές συνθήκες ή από επιζωτίες ε, που ξεσπάνε. Ε, θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να αντιδρούμε άμεσα σε περίπτωση που ανακύπτουν τέτοιες κρίσεις, θεομηνίε, ε, ζωνώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον κύριο Βιώτη, αλλά και τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση γιατί σίγουρα με τις παρεμβάσεις τους εμπλουτίζουν και τη δική μου ε, γνωμοδότηση. Στα τέλη Απριλίου είχε λήξει η διορία για τις τροπολογίες, κατατέθηκα 44 τροπολογίες, μια και έχει λήξει προθεσμία, δεν μπορώ να δεχτώ άλλες τροπολογίες, αλλά οι ιδέες που παρουσιάστηκαν στη συζήτηση ε, θα με βοηθήσουν και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο που θα εξυπηρετεί το σκοπό μας, που είναι η προάσπιση των αγροτών μας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι στις εκλογικές μας περιφέρειες κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και πολύ καλοπροαίρετα όλοι με καλή βούληση, είναι αναφυσβήτητο, δεν ε, αμφιβάλλω για την καλή βούληση που έχουμε και την καλή πρόθεσή μας να προσπίσουμε τους ε, γιώργους μας. Ανέκυψε το ζήτημα του ρωσικού εμπάργου και φαίνεται ότι υπάρχει επιφύλαξη για την παράταση ή τη διέμβριση των ενισχύσεων. Εγώ την Παρασκευή θα πάω σε μια συνάντηση με αγρότες ε, στη γενέτειρά μου, στη Μούρσια τι να τους πω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη συνέχιση ή την ενίσχυση των κονδυλίων για να αντιμετωπιστεί το ρωσικό εμπάργο. Ποιον θα πείσω, ποιον θα καθησυχάσω με τέτοια βεβαιότητα. Είναι αλήθεια βέβαια ότι αυτό δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό του 2019 και τη γεωργία. Αλλά αν κάπου κολλήσουν οι διαπραγματεύσεις ή αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις του Brexit, τι θα γίνει. Θα βρεθούμε μετέωροι και δεν έλαβα συγκεκριμένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, για να μην μιλήσουμε για τη γεωργία. Η γεωργία εκφύσεως πάντα περιβάλλεται από αβεβαιότητα. Τώρα στην γνωστή αβεβαιότητα της γεωργίας λόγω καιρικών και άλλων συνθήκων να προσθέσουμε και την πολιτική αβεβαιότητα που δεν μπορούμε ακόμη να καλύψουμε γιατί δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει μια δεχόμενη αποτυχία των διαπραγματεύσεων του Brexit. Τι θα πούμε στους Γιώργους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σίσο, ευχαριστούμε κύριε Βιώτη. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης. Τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων έγινε η παρουσίαση της οδηγίας ε, για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών από τον Επίτροπο. Ε, έχουν μακροχρόνια πορεία αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τις γνωρίζουμε και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και πολλές χώρες μέλη θέσπισαν ε, τα δικά τους μέτρα, αλλά έχουμε ενιαία αγορά, γι' αυτό χρειάζονται πανευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Πάντως η Σλοβακή Προεδρία ε, θέσπισε σε ειδική ομάδα για την ανάλυση αυτού του θέματος με πρόεδρο τον Επίτροπο Χόγκαν. Έκανε πολλά η Σλοβακή Προεδρία για το θέμα αυτό. Και έχουμε και την έκθεση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. στην οποία συμμετείχε εκ μέρους μας ε, και πρόσφερε πολλά η κυρία Μαγκίνες. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο στον εισηγητή μας για το θέμα αυτό, στον κύριο Δεκάστρο καλωσορίζοντας και τους ε, εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα είναι ε, πολυμελής η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι σχετικά συνήθιστο. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έτσι είστε περισσότεροι που ακούτε τις ε, παρεμβάσεις και τις απόψεις των μελών της Επιτροπής Γεωργίας. Κύριε Δεκάστρο, έχετε το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από τα συναδέλφους ε, λιγάκι να με προσέξουν. Πρώτα απ' όλα, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ότι ε, πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση που είναι το αποτέλεσμα δεκαετούς ε, προετοιμασίας και εδώ στο Κοινοβούλιο όσο και στην Επιτροπή. Μετά τον καψέ από τις προτάσεις της Task Force για τις αγροτικές αγορές και αγορές τροφίμων. Όπως ξέρετε η Task Force ε, έλαβε πάρα πολλά κίνητρα κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον κανονισμό Omnibus. Η οδηγία λοιπόν αυτή είναι να την καταστήσουμε ακόμα πιο φιλόδοξη. Να έχουμε όμως ε, κατά νου ότι είναι πολύ ευαίσθητες ε, οι ισορροπίες τις οποίες υπερισχύουν ε, οι δικές τους οδηγίες, υπάρχει ένα επίπεδο εγγύησης. Να βελτιωθεί η αντιμετώπιση παράτυπων διαδικασιών ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διευρύνουν αυτόν τον κατάλογο και θέλω να εκφράσω και δύο απόψεις ε, για το πρόγραμμα εργασίας. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε αμελητή. Αμελητή λοιπόν οι εργασίες για να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας της 10 Ιουλίου την έκθεση να το παστέ να συγκεντρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες προτάσεις από τις διάφορες ομάδες. Και αυτό για να αποφύγουμε μετά να έχουμε να κάνουμε με εκατοντάδες ε, τροπολογίες. Ε, θέλω να περιοριστούν οι τροπολογίες. Ε, όπως σας είπα από την Επιτροπή Γεωργίας, αυτό ήδη μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο και πρώτη-δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα πάμε για ψηφοφορία στην Ολομέλεια με εντολή διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή έχει ήδη κάνει δύο συναντήσεις, ε, έχει ήδη γίνει αρκετή δουλειά και την θητεία του Κοινοβουλίου να μπορέσουμε να καταλήξουμε φινάδελφοι και καταλήγω για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο μας είναι σημαντικό να κερδίσουμε μία μάχη που μένεται και εδώ απευθύνομαι στον πρόεδρο και τη γραμματεία. Γιατί όπως γνωρίζετε η Επιτροπή ΙΜΚΟ διεκδικεί, άρα δηλαδή είναι σαφής, ε, δεν μπορεί να δοθεί σε αυτή την Επιτροπή, την ΙΜΚΟ. Παρόλα αυτά εγώ ίσως ε, προκαλώντας τους ε, της Επιτροπής ΙΜΚΟ, αλλά δεν γίνεται σε αυτήν την θητεία. Άρα υπάρχουν νομικοί και πολιτικοί λόγοι που μας οδηγούν να περιοριστούν οι τροπολογίες. Να έχουμε μία έκθεση που θα εκφράζει όλες τις απόψεις και η έκθεση αυτή. Και έγινε διάλογος μεταξύ των γραμματιών των δύο επιτροπών. Εμείς ετοιμάσαμε πολύ βάσιμα επιχειρήματα που θα μας επιτρέψουν να διαφυλάξουμε την αρμοδιότητα για αυτό το θέμα οι σκιώδεις για δύο λεπτά ο καθένας και οι υπόλοιποι για 1,5 λεπτό. Κυρία Μαγκίνες, που είχε λάβει μέρο και στην προηγούμενη εκδοχή αυτής τη έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε. Πριν το τέλο της θητείας μας αυτό όμως απαιτεί πειθαρχία από εμάς για να παραμείνουμε εντό των αρμοδιών. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια διαμάχη μεταξύ των επιτροπών. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας πει ο πρόεδρος πότε θα ξεκαθαρίσει. Τι υπάρχει το άρθρο 53, 54 μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να το δούνε και το χρονοδιάγραμμα και το τι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. E, myśmy e, Εμείς ε, ε, δώσαμε τα επιχειρήματά μας στον πρόεδρο της διάσκεψης ε, των πρόεδρων. Μιλήσαμε για, το, για τις διορίες, για την αρμοδιότητα, για το χρονοδιάγραμμα. Θέσαμε όλα αυτά τα ζητήματα και μπορούμε να στείλουμε στους ενδιαφερόμενους τη σχετική επιστολή που στείλαμε στον πρόεδρο της διάσκεψης των πρόεδρων. Ίσως ε, μπορούν να το εμπλουτίσουν και με άλλα επιχειρήματα, παρόλο που τα έχουμε στείλει ήδη, αλλά συνεχίζεται η συζήτηση τους ή άλλως. Η κυρία Μακιντάιρ. Uh, thank you, Chair. Um, Μα αυτά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Γεωργίας. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό. Και νομίζω και διότι η αρμοδιότητα ότι είναι πολύ σημαντικό να περάσει αυτή η νομοθετική πράξη. Εγώ το επιθυμώ αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Γιατί θέλω να είμαι ήδη κατά το παρελθόν δουλειά και λήφθη υπόψη στην διατύπωση της πρότασης που μας κατατέθηκε. Προσβλέπω στο να συνεργαστώ λοιπόν μια καταπληκτική βάση και νομίζω υπάρχει και κάτι άλλο με το οποίο και θα κλείσω. Το 94% της... αυτό και μόνο δείχνει πόσο σημαντικό είναι το όλο θέμα. Η κυρία Χόιμπους. Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα είναι επίσης ε, σημαντικό και θέλω να υποστηρίξω τον κύριο Δεκάστρο στο ότι πρέπει να παραμείνει θέμα της Επιτροπής μας και να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο δεν ανέφερε η Κομισιόν. Οι σχέσεις ε, δηλαδή του εμπορίου με την ε, δική μας την, ε, και τους, αυτούς οι οποίοι επεξεργάζονται τα τρόφιμα, να δούμε δηλαδή ακριβώς ποια είναι η σχέση γεωργών με αυτούς οι οποίοι δίνουν, δίνουν τα προϊόντα τους στις βιομηχανίες που τα επεξεργάζονται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για μια υπόθεση και ένα θέμα της Επιτροπής Γεωργίας. Βεβαίως ε, μπορεί και να διευρυνθεί η έκθεση, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει από την μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς στον τομέα των τροφίμων και δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Κλείσουμε. Ο κύριος Τσούλο. Grazie, Presidente στους πολίτες αλλά και στην ε, ε, κοινή αγορά. Γνωρίζουμε ότι η παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ε, Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από την Επιτροπή. Σημείωσα ότι δεν υπάρχει κάποιος ορισμός ε, για τις αθέμητες εμπειρίες ε, παράνομες πράξεις και να εντάξουμε αυτή στον ορισμό. Ένα δεύτερο που θέλω να είναι το εξή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι λιγάκι επικίνδυνο, γιατί δεν νομίζω ότι θέλουμε να υπάρχει οδός διαφυγής ε, για τις πολυεθνικές. Εμείς θα θέλαμε οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να ε, προστατεύονται από παράτυπες και παράνομες πρακτικές, από οπουδήποτε και αν έρχονται αυτές και τεύση να είναι προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ θα ήθελα να υιοθετήσουμε αυτή την πρακτική ε, δηλαδή να δώσουμε την αρμοδιότητα ε, στον ε, προμηθευτή του προϊόντος και όχι να επιβάλλουμε Μπορείτε να μιλάτε ελληνικά, αλλά πρέπει να ακούτε μία άλλη γλώσσα. Χαίρετε. Olen myös ehdottomasti sitä mieltä, että tämä kuuluu akralla. On elintarvikeketjun lainsäädäntöä, antaa vahvan selkänojan myöskin EU-lainsäädännölle